κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με τρόπο δίκαιο και ισότιμο. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και αντίστοιχη ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα στρατηγική εσωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων. Κύριε Επίτροπε, καλησπέρα σας. Ο συντάκτης. Το λόγο έχει για πέντε λεπτά ο κύριος Λόπες Αγγελάρ. Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη στρατηγική εσωτερική ασφάλεια που εγκρίθηκε στο πρώτο εξάμεινο του 2010 επί Ισπανική Προεδρία, θυμάστε αρχές λοιπόν και κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να διέπουν σε σχέση με τη στρατηγική και τις απειλές στην Ευρώπη. Είναι ε, μέτρο κλειδί του προγράμματος της Σοχόλμης και εκπονείται τώρα ένα σχέδιο για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 67 του, ε, της Συνθήκης Λισαβόνας και μιλά για τις πιο κρίσιμες απειλές προς την κοινή μας ασφάλεια όπου μπορεί και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει προσθέμενη αξία ε, να σταματήσουν τα οργανωμένα εγκλήματα από δίκτυα ή τρομοκρατία, να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια, να ενισχυθεί η προστασία των εσωτερικών συνόρων και να αυξηθεί η πολιτική προστασία απέναντι σε θεομηνίες. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Πάρα πολύ από το 2010 είναι τεράστιες οι προκλήσεις και νέες οι απειλές και χρειάζονται διαφοροποιημένες πολιτικές απαντήσεις για να γνωρίζει και να ενημερώνεται η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, συνεργάζεται με την Ευρωπόλ, με το σημερινό ε, συντονιστή κατά της τρομοκρατίας, τον κύριο Ντεκέρχοφ και συζητάει για τις τελευταίες τάσεις στην εγκληματικότητα και ε, την τρομοκρατία και με το Διευθυντή της Ευρωπόλ συζητούμε για την έκθεση για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και την ε, αντίστοιχη έκθεση αξιολόγηση που αποτέλεσε τη βάση για να αποφασίσει τον Ιούνιο το Συμβούλιο τις νέες προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, την επόμενη τετραετία. Στο ψήφισμα της Επιτροπής Ελευθεριών υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις για τις νέες προτεραιότητες. Δηλαδή, συγκεκριμένες συστάσεις ακριβώς για τις προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων, ε, το λαθρεμπόριο όπλων, αυτά είναι στρατηγικές προτεραιότητες. Και με τον κύριο Ντεκέρχοφ που είναι συντονιστής κατά της τρομοκρατίας συζητήσαμε την έκθεση για τη νέα κατάσταση στην τρομοκρατία. Η λεγόμενη ε, μοναχική λύκη. Είναι νέα μορφή τρομοκρατίας αυτή, με μονομένα άτομα που δρούν εξάρτητα. Συνεργαζόμαστε με την ε, ε, προσωρινή Επιτροπή ΚΡΙΜ, που εστιάζει κυρίως ε, στο ξέπλυμα χρήματος, στη διαφθορά και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε. Η Επιτροπή χρειάζεται να αξιολογεί και να ενημερώνει την κατάσταση αυτή και το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί με ένα κριτικό μάτι την κατάσταση και να θέτει τις προτεραιότητες. Το κάναμε πέρσι με εισηγήτρια την κυρία Μπορσελίνο και πάλι και σήμερα είναι η δεύτερη έκθεση εφαρμογής, τη συζητούμε και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο τράφικινγκ, στη διακίνηση ανθρώπων, ε, στο κυβερνοέγκλημα, ε, στην τρομοκρατία, στην ιδιαίτερη βία, το οργανωμένο έγκλημα παραμένει εσωτερική απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο κατά της ασφάλειας, αλλά και κατά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και ε, είναι και θέμα που αφορά την οικονομική κρίση. Και μιλούμε για την τέταρτη οδηγία κατά του ξεπλήματος, για την οδηγία την προστασία των... Ε, ε, ε οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Είναι περίφημη οδηγία που έχω την τιμή να είμαι προ, Επίσης, ε, η Επιτροπή Ελευθεριών θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προλαμβάνει τις εξελίξεις και να δραστηριοποιείται κατά του εγκλήματος ε, και ιδιαίτερα σε θέματα ε, περιβάλλοντος, λάθρεμπορίου, βελτίωση του ελέγχου των συνόρων και οι λεγόμενες κρίσιμες υποδομές. Επίσης υπάρχει και μια δικαστική διάσταση, να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός δικαστικός ε, ε, πολιτισμός και να ξέρουμε και τα δικαιώματα, τα δικονομικά. Αλλά με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Σαββόνα συμμετέχει όσο ποτέ το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Λίμπε στο δημοκρατικό έλεγχο αυτής της πολιτικής και της εφαρμογής της. Ευρωπαϊκό χάρτης λέμε θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πλέον δεσμευτικό. και η Επιτροπή ΛΥΠΕ θα πρέπει να ενημερώνεται και να δρά σχετικά ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν προετοιμάσει τη νέα στρατηγική για το 2014 θα πρέπει να συνεργάζεται με τη δική μας Επιτροπή όπου θα έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τέλος θέλω να σας πω ότι η στρατηγική εσωτερική ασφαλείας συχνά είναι αρμοδιότητα κρατών μελών. Γι' αυτό θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συνεργάζεται στενά με τα Εθνικά Κοινοβούλια, πράγμα που πράττουμε εμεί κάθε έξι μήνε. Στο ψήφισμα της Επιτροπής Ελευθεριών επαναλαμβάνουμε αυτή την ιδέα να έχουμε κοινέ ε, ε, κοινοβουλευτικές διασκέψεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε ένα κύκλο κοινοβουλευτικό στην Ευρώπη και να συμπεριλαμβάνεται και η έκθεση αυτή για τη στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Χωάν Φερνάντο. Το λόγο έχει ο Επίτροπος, κύριος Άντορ, για να απαντήσει στην προφορική ερώτηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Η στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας εφαρμόζει ένα τμήμα του προγράμματος του Στοκχόλμης, ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας του πολίτη. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στην περίοδο μετά τη Στοκχόλμη θα πρέπει να τοποθετηθούμε απόλυτα στο νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Λισαβόνας και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό, τον ε, ευπρόσδεκτο ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην νομοθετική διαδικασία και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Γίνεται προβληματισμό όσον αφορά την περίοδο μετά Στοκχόλμη και σκοπεύουμε να κάνουμε ανακοίνωση όσον αφορά τι πολιτικέ εσωτερική πολιτική το Μάρτιο, τον επόμενο χρόνο. Πράγμα το οποίο θα συμβαδίσει με την ανακοίνωση για τι μελλοντικέ προτεραιότητε περί δικαιοσύνη. Η Κομισιόν πρέπει να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις και συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 22 Μαΐου 2012 για την ε, εσωτερική πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δεύτερη δηλαδή έκθεση για το ISS και αυτό θα περιλαμβάνεται και στην τρίτη ε, έκθεση εφαρμογής για την ε, ε, στρατηγική εσωτερική ασφάλειας. Έχει υπάρξει πρόοδος για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Τα μεμονωμένα σημεία του ψηφίσματος λαμβάνονται επίσης υπόψη σε σχέση με τα σχετικές ε, ε, θεματικές της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Θα μπούμε τώρα στους συναδέλφους που θα μιλήσουν εξ ονόματος των πολιτικών τους ομάδων. Για δύο λεπτά ο κύριος Κούρια εξ του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Επίτροπο όσο και το δικό μας ε, εισηγητή και Πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, Λόμπες Αγγιλάρ, για αυτή την ερώτηση, για αυτή την έκθεση. Ε, λέω, ψηφίσει το Κοινοβούλιο για κάποιε πτυχές τι οποίε ε, έχουμε θεωρήσει πολύ σημαντικέ. Καταρχήν βελτίωση τη δυνατότητα ανάλυση των φυσικών κινδύνων γιατί πιστεύουμε κυρίω σε φάσει δύσκολε όπω ε, οι πλημμύρες, ε, οι σεισμοί. Οι Ευρωπαίοι πολίτε θα πρέπει να δουν μια Ευρώπη έτοιμη να δώσει βοήθεια και άμεση στήριξη. Συχνά όταν κάποια κρατημέλη βρέθηκαν συγκλονισμένα από φυσικέ καταστροφέ. η απάντησή μα δεν ήταν άμεση ούτε πλήρη. και η αλληλεγγύη θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία της Ένωσης. Δεύτερον, έχουμε υπογραμμίσει το ρόλο του θέματος των εξωτερικών ε, συνόρων που είναι απαραίτητα για την εσωτερική μας ασφάλεια. Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση των ε, ε, μεταναστευτικών ροών έτσι ώστε ο μεγάλος αριθμός μεταναστών να μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Έχουν δικαίωμα οι μετανάστες σε ανθρώπινη και δημοκρατική υποδοχή όταν όμως δυσανάλογα μεγάλοι αριθμοί φτάνουν δημιουργούνται προβλήματα προβλήματα, δυσκολίες ε, τόσο για αυτού που φτάνουν όσο και για όσους τους υποδέχονται. Να δεν υπάρχει δηλαδή ε, ρύθμιση, υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο στου πολίτες και αυξάνεται η ανασφάλεια και αυτό θα πρέπει να επηρεάσει τις δικές μας ε, ρυθμίσεις. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία. Υπάρχουν ακόμα πολλές, ε, πολλά περιστατικά βία εναντίον γυναικών και παιδιών και για μας αυτά ενδιαφέρουν ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση της εσωτερικής ασφάλειας, αν και κάποιοι υπέβαλαν ε, τροπολογίες για να ακυρώσουν το κομμάτι που αφορά την καταπολέμηση της παιδοφιλίας. Υπάρχουν ε, τμήματα ε, τα οποία δεν μας πείθουν απόλυτα. Το πιο σημαντικό όμως είναι να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια συνολική στρατηγική που θα δίνει εγγύησεις και ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό άλλωστε βρισκόμαστε εδώ. Ευχαριστούμε. Εξ σοσιαλιστών έχει τώρα για δύο λεπτά το λόγο ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη για τους περισσότερους πολίτες της δεν είναι μόνο οικονομικό εγχείρημα με ενιαία αγορά ε, περιμένουν κοινωνική συνοχή και ελευθερία και ασφάλεια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα προς ένα χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Εξούσου σημαντικό και πολύ μάλιστα είναι και η κοινοτική διάσταση ε, αυτής και η ίση συμμετοχή και των τριών θεσμικών οργάνων. Κομισιόν, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου. Συχνά μου λείπει η βούληση των υπολείπων να λαμβάνεται ε, όπως που αναλογεί υπόψη το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό τα πέντε σημεία της στρατηγικής αυτής θα είχαν εμπλουτιστεί εάν ήταν προσανατολισμένα περισσότερο ε, στα μελήματα και στις ανησυχίες των πολιτών. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, είναι υπαρξιακό το θέμα της ασφάλειας αλλά δεν θέλουν να χάσουν και την ελευθερία τους. Η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, είναι βασική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό η κριτική μας είναι κάπως και κάτι επικοδομητικό. Και πολύ σημαντικό επίσης είναι το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου των ευρωπαϊκών οργανισμών που δραστηριοποιούνται εδώ. Πολλά μέτρα λαμβάνονται διστακτικά και η νομοθετική πράξη για την Ευρωπόλ μπορεί να ολοκληρωθεί κατά την παρούσα θητεία. Και η συμπερίληψη των εθνικών κοινοβουλίων θα μπορούσε να γίνει με τρόπο πιο ενεργό και δραστήριο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την οδηγία για την επεξεργασία των δεδομένων από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Θα ήταν ένα σημαντικό μήνυμα για σύγχρονη ε, νομοθεσία για το συγκερασμό της ασφάλειας με την ελευθερία. Ευχαριστώ Γιώζεφ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Άλμπρεχτ, τον οποίο δεν βλέπω στην αίθουσα, αλλά μπορεί να μην είναι στο έδρανό του και να είναι αλλού. Κανονικά θα έπρεπε να μιλήσει εξ ονόματο των Πρασίνων, αλλά απουσιάζει όντω. Αν έρθει αργότερα θα του δώσουμε το λόγο. Από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, για ένα λεπτό, ο κύριο Κέρχοπ. Uh, uh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, υποστηρίζω ε, πλήρως την ανάγκη ε, να θεσπίσουμε ε, μια στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια, την ασφάλεια των συνόρων, την ασφάλεια των πολιτών και τη δράση της Ένωσης στον τομέα αυτό. Έχω, υποστηρίζω το έργο της Ευρωπόλ και την ανάγκη καλής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών για τα εγκλήματα και την τρομοκρατία. Έχουμε τομείς που δεν έχουν προτάσεις για λύση. Βεβαίως ε, η προστασία και τα, ε, και τα δικαιώματα τα ατομικά ίσως ε, έρχονται σε αντιπαράθεση. Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Ε, ε, βεβαίως ο εισηγητής ε, είναι ένας καλός άνθρωπος και πρέπει να υποστηρίξουμε ε, τις προσπάθειές τους. Θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική συνεκτική και χρήσιμη. Μην έχουμε μικτά μηνύματα σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ πολύ για να ολοκληρώσουμε τους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Κορνέλια Έρνστ εξ ονόματος της Συνοτικής Αριστεράς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια και εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να έχουν στρατηγική εσωτερική ασφαλείας. Και υποστηρίζουμε εδώ τον εισηγητή, δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Για μας το πιο αποφασιστικό ζήτημα είναι ποια είναι η σχέση ασφάλειας με την ελευθερία των πολιτών και αν έχει σταθμιστεί επαρκώς. Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς αυτή η σχέση και ειλικρινά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούω κούφια λόγια και μόνο. Δεν μπορούμε με κατασταλτικές στρατηγικές και καταπιεστικές να στραγγαλίζουμε τους πολίτες κράτος δικαίου σημαίνει ότι το κράτος υπάρχει για τους πολίτες και όχι πολίτες για το κράτος. Και αυτό θα πρέπει να είναι και στόχος αλλά και κατευθυντήρια γραμμή της στρατηγικής. Ξέρετε, εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου κατά πόσο με τις στρατηγικές μέχρι σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε. Με τις στρατηγικές που έχουμε σκεφτεί δηλαδή. Γιατί ξέρουμε ποια είναι τα γεγονότα και το σκάνδαλο με την NSA. Και σας ερωτώ τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σταματήσει αυτό το φακέλωμα και η κατασκοπία εκατομμυρίων πολιτών. Είναι κρατικά οργανωμένη εγκληματικότητα αυτό στην ουσία. Τι κάνετε για να εξασφαλίσετε την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των πολιτών που τόσο ωραία μας τα περιγράφετε. Είναι σκανδαλώδης αυτή η κατασκοπία κατά των πολιτών μειώνεται και το κατόφλι της υποψίας ε, και αυτό είναι και εις βάρος της ε, κατασκοπίας και της τρομοκρατίας και της καταπολέμησης. Αυτά δεν είναι λύση ασφαλείας, είναι πρόβλημα για την ασφάλεια και θα πρέπει να τα καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ. Έχουμε ορισμένου μεμονωμένου τώρα βουλευτέ που μιλούν ε, ατομικά και πρώτα για δύο λεπτά ο κύριο Αγουστίν Δία Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ επικαιρή και εύστοχη η ερώτηση του κύριου Λόπες Αγγιλάρ. Θα ήθελα να σας πω κάποιες προτεραιότητες που θεωρώ σημαντικές και που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη για τη μελλοντική εφαρμογή της ε, στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Πρώτον, ο πολύ σημαντικός ρόλος των ευρωπαϊκών οργανισμών για να φτάνουμε στους στόχους μας σε θέματα που μας απασχολούν. Η ιδιαίτερη Ευρωπόλ είναι πολύ σημαντική. Στις 27 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε νομοθετική πρόταση και είμαι συγητής για αυτή. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, επανειλημμένη άποψη που έχουν εκφράσει ε, τα ε, κόμματα, πολιτικές ομάδες δηλαδή και τα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο Τζάι 7 Ιουνίου. επαναλαμβάνω την αντίθεσή μου πιθανής ε, σύνδεξης και συνένωσης Ευρωπόλ και ΣΕΠΟΛ. Έχουν ξεχωριστή δουλειά διακριτό ρόλο και θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν. Γι' αυτό παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα να καταθέσει την πρόταση κανονισμού που αφορά μόνο ε, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, τη ΣΕΠΟΛ δηλαδή. Και θα πρέπει η Κομισιόν να εξετάσει τις προτεραιότητες του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ η Ισπανία στις επιχειρήσεις αυτές, θα συμμετάσχει σε όλες. Θα είναι επικεφαλής σε δύο και μόνη της και σε ε, δύο μαζί με κάποιους άλλους. κατά πολέμηση ε, κοκαίνης, ε, ηρωίνης, του λαθρεπορίου και όπλων. Ε, παραμένει εν ζωή η τρομοκρατία και έχουμε διάφορες εκφάσεις και θα ήθελα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ριζοσπαστικοποίηση των μαχητών και των λεγόμενων μοναχικών λύκων μεμονωμένων τρομοκρατών. Και τέλος, θα ήθελα να μιλήσω και για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να υπάρξουν και απαραίτητοι ε, πόροι ε, στον άξονα 3 που εξαρτάται από την Ευρωπόλ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και δύο λεπτά τώρα ο συνάδελφος Παπα-Νικολάου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, τον κύριο Λόπεζ Αγγιλάρ, για την σημερινή πρωτοβουλία να έχουμε αυτή την σημαντική συζήτηση. Πράγματι, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, εμπεριέχει πολύ σημαντικά δεδομένα, κάποια από τα οποία καταφέραμε να αξιοποιήσουμε ε, τα χρόνια που πέρασαν. Και στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και έχουμε πρόοδο. Διερωτάται όμως κανείς, φτάσαμε στο επίπεδο εκείνο να πιάσουμε τους στόχους του προγράμματος Στοχόλμης. Νομίζω η απάντηση στο ερώτημα αυτό, και απευθύνομαι στον κύριο Επίτροπο που ανέφερε το πρόγραμμα, είναι όχι. Δεν καταφέραμε σήμερα να ε, φτάσουμε στα επίπεδα της αλληλεγγύης που το ίδιο το πρόγραμμα προβλέπει και η ίδια η συνθήκη προβλέπει στη δίκαιη κατανομή των βαρών σε συγκεκριμένους από τους πυλώνες που περιγράφει και το πρόγραμμα για την εσωτερική μας ασφάλεια. Κουβεντιάζαμε στην Ολομέλεια σήμερα, πριν από αυτή τη συζήτηση, για τις προκλήσεις σε σχέση με την κατάσταση στη Συρία και την Αίγυπτο ένα από τα ζητήματα που κουβεντιάσαμε είναι οι μεγάλες ροές ετούντων άσυλο που θα φτάσουν στα εξωτερικά σύνορα της ένωσης και θέλω να δώσω έμφαση ακριβώς σε αυτό το σημείο. για να έχουμε εσωτερική ασφάλεια πρέπει να έχουμε και ολοκληρωμένη προστασία των εξωτερικών μας συνόρων και αναμένουμε βεβαίως πολλά και από τη νέα πρόταση που σύντομα ελπίζουμε θα ψηφιστεί για τη eurosur. Ε, είμαστε στο επίπεδο να πιστεύουμε σήμερα ότι υπάρχει δίκαιη κατανομή των βαρών και πλήρης και πραγματική αλληλεγγύη στο ζήτημα αυτό ε, και συνεργασία με τα κράτη μέλη. η απάντηση δυστυχώς δεν είναι θετική. δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο κράτη μέλη δυσανάλογα να επιβαρύνονται σε σχέση με κάποια άλλα. αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την ανάπτυξη του ρατσισμού της ξενοφοβίας σε πολλές χώρες το, το ζούμε καθημερινά το καταλαβαίνουμε να ενισχύεται ε, όσο περνάει ο καιρός και βεβαίω αυτό συνδέεται άμεσα και με τον εξτρεμισμό. καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά τελικά έχουν ως αποτέλεσμα και η ίδια η εσωτερική μας ασφάλεια να μην είναι αυτή που θα θέλαμε. Βεβαίως έχουμε πολλά να κάνουμε, βεβαίως έχουμε επιτύχει σημαντικά βήματα, είναι όμως μεγάλες οι προκλήσεις για τη συνέχεια και αναμένουμε στις επόμενες προτάσεις της Επιτροπής συγκεκριμένα ε, βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Για δύο λεπτά ο κύριος Γιακολίνο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνθήκη της Λισαβόνας καθόρισε και έδωσε αυξανόμενες ευθύνες στο Ευρωκοινοβούλιο και στην διακυβέρνηση αυτό που αποκαλούμε στρατηγική ιστορικής ασφάλειας. Η πρόταση του Πρόεδρου δεν μπορεί παρά να στηριχθεί επειδή στηρίζεται σε αυτές που είναι οι προτεραιότητες παρέμβασης μιας πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ολοκληρωμένα να ασκήσει και σε συμφωνία και συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει αμφιβολία, για παράδειγμα, ότι το θέμα που αφορά την ε, ασφάλεια την ε, ε, ψηφιακή είναι πολύ σημαντικό θέμα. Μπορεί να δοθεί δε στήριξη από την αρμόδια υπηρεσία που πρόσφατα δημιουργήθηκε προς την Ευρωπόλ, καθώς και να γίνουν δράσεις διαρκώς υπέρ της διατήρησης ε, της ιδιωτικής ε, σφαίρας, της προστασίας μάλλον της ιδιωτικής ε, σφαίρας. Επίσης, ενέργειες κατά της θερμοκρατίας, της μαφίας, του οργανωμένου εγκλήματος. Γι' αυτά όλα χρειάζεται έκτακτη συνεργασία δικαστική και αστυνομική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη καθώς και ένα ανανεωμένο πρόγραμμα σύνδεση με τις τρίτες χώρες που θα συλλέγονται οι πληροφορίες προστατεύοντας όμως τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα. Κατά τη της τρομοκρατίας, πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, για το οποίο είμαι και εισηγητή και για την ανακύκλωση βρώμικου χρήματος. Μια ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να δώσει μεγάλα και σπουδαία αποτελέσματα. Τώρα, μετανάστευση και κινητικότητα. Πρέπει και εκεί να συνεργαστούμε πιο στενά με τις χώρες που εκτίθενται περισσότερο σε πίεση μεταναστευτική διαρκώς στα θαλάσσια μας σύνορα αλλά και στα επίγεια σύνορα να μπορέσουμε να δώσουμε ευκαιρίες ε, απασχόλησης στους νέους μας. Η Συρία και η Αίγυπτος προφανώς απέδειξαν την αποτυχία της Αραβικής Άνοιξης και όχι μόνο εκείνης, ας πούμε στα κρατημέλη να ενεργήσουν ε, υπεύθυνα και με αλληλεγγύη. Χρειάζεται ένα μια νέα όθηση, Πρόεδρε, από τη Βαλτική ως την Μεσόγειο. Μια ισχυρή συνεργασία που θα μπορέσει να εγγυηθεί τέτοια αποτελέσματα, αυτά που αναμένουν οι, τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Μια αύξηση της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Τελευταία ομιλήτρια σε αυτό το γύρο είναι η κυρία Χιμένες Μπεσερίλ για δύο λεπτά επίσης. Τερέσα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από 12 χρόνια τέτοια μέρα, θυμάστε τι έγινε, μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση της ιστορίας Περίπου 3.000 ήταν οι νεκροί και 6.000 οι τραυματίε στην Αμερική την 11η Σεπτεμβρίου. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμή σε όλα τα θύματα τη τρομοκρατία εντό και εκτό τη Ευρώπη. Έχουμε ένα χρέο απέναντι σε όλου αυτού που έχασαν τη ζωή του γιατί εκπροσωπούσαν αξίε στι οποίε εμεί είμαστε προσιλωμένοι, βασικά την ελευθερία. Το θέμα που μα απασχολεί σήμερα έχει να κάνει με τη στρατηγική εσωτερική ασφαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ω βασικό στόχο με τη σειρά τη, προστασία της ζωής των πολιτών. Χαίρομαι λοιπόν που η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική αυτή θεωρεί την τρομοκρατία ως προτεραιότητα. Εξακολουθεί να την έχει στο κέντρο της, ε, την πρόληψη και την καταπολέμηση της ε, ρίζος Σύμφωνα με την Ευρωπόλ η απειλή από την τρομοκρατία έχει πολλές εκφάσεις από την Αλκάιδα μέχρι τους αποσχιστές τρομοκράτες και το άρθρο 12 της πρώτας ψηφίσματος ζητεί να διερευνηθούν ε, οι ε, βίες ε, εκφάσεις της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και εγώ αναρωτιέμαι η ακροαριστερά δεν έχει βίες εκφάνσεις και ο σεχταρισμός είναι εις βάρον όλων και η τρομοκρατία απαντά σε μία και μόνη ιδεολογία του φόβου του τρόμου και του πόνου. Θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι με καλύτερη εκπαίδευση των ειδικών στην αντιτρομοκρατία, με μεγαλύτερη δυνατότητα απόκρισης από πλευράς των πολιτών. Να ακούμε τις μαρτυρίες των μαρτύρων ακριβώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχυθεί η κατηγορία και η καταδίκη για τρομοκρατία. Το 2015-2019 στην επόμενη περίοδο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα μελήματα και στις προσδοκίες των πολιτών που θέλουν να ζουν σε ασφάλεια και ελευθερία. Εγώ είμαι προσιλωμένη σε αυτό και είμαι βέβαιο ότι και όλο το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Τερέσα. Μία συνάδελφο ζήτησε το λόγο στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑΗ και είναι η κυρία Ρόιτοβα και τη δίνουμε αμέσω το λόγο. Ξέρετε ότι έχετε ένα λεπτό σε αυτή τη διαδικασία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βεβαίως η υλοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος είναι βασικές προκλήσεις που μας απασχολούν σήμερα. Ε, χαιρετίζω νέα νομοθεσία ε, για ε, την κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματος και αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα εκρηκτικά. Αλλά το σημαντικότερο πίτευμα που είναι η εκπαίδευση, η αντιτρομοκρατική που ε, κατά των ε, φανατικών ομάδων των φονταμανταλιστών. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την ε, συνεργασία των κέντρων κατά των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, κέντρα τα οποία θα μπορούν να αποτελέσουν πλατφόρμα για ανταλλαγή εμπειριών. Ευχαριστώ. Για να κλείσει τη συζήτηση, το λόγο έχει ο Επίτροπος που θα απαντήσει και στην ερώτηση και τα σχόλια που του έγιναν από όλους τους συναδέλφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη και κυρίως τον κύριο Λόπεζ Αγγιλάρ ε, για αυτήν ε, την πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση για την στρατηγική εσωτερική ασφάλειας με συγκεκριμένες προτάσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Παπα-Νικολάου ότι η εσωτερική ασφάλεια απαιτεί πλήρη συνεργασία και περισσότερη αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Μερικά από τα θέματα που αναφέρθηκαν στη συζήτηση θα απαιτήσουν ίσως ενδελεχή αξιολόγηση των διαφόρων πρακτικών και συμβάντων αλλά νομίζω ότι η συζήτηση αυτή ήταν ε, σημαντική για την ε, εφαρμογή, υλοποίηση του προγράμματος της Στοχόλμης για την ικανοποιητική εσωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έχουμε λάβει ένα πρόταση, πρόταση ψηφίσματος, πρόταση ψηφίσματος. Θυμίζω σε όλους σας ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τώρα η κατάσταση είναι λίγο ε, άβολη, πώς να το πω. Το επόμενο θέμα στην ημερησία δέταξη που είναι και το τελευταίο, σε αυτή την πολύ μακρά ημέρα, είναι μια προφορική ερώτηση μια συναδέλφου που παρευρισκόταν εδώ στη συζήτηση για πολύ χρόνο, αλλά τώρα απουσιάζει.